Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι έχουμε απαρτία για να ξεκινήσουμε. Άρχεται λοιπόν η συνεδρίασή μας. Δεν βλέπω αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη, οπότε μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ε, δεν έχει πολλά σημεία. αλλά το εύρος της συζήτηση θα είναι ευρύ, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα. Έχουμε διερμηνία σε 19 γλώσσες, με εξαίρεση φιλανδικά, ιστανικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και ιρλανδικά και ελτικά. Όπως ξέρετε, είναι εκτακτή η συνεδρία της Επιτροπής και το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αφορά την ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο για την κατάσταση των αγορών γεωργικών προϊόντων. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν που ήρθε για ανταλλαγή απόψεων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθατε κύριε Επίτροπε, ώστε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Και μάλιστα ε, βρίσκεται παρόν είναι παρόν στη συνεδρίαση και ο κύριος Αρτουή, ο πρόεδρος τη Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον ευχαριστώ και καλωσορίζω. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και συνήθως η συζήτηση πολύ σημαντικών θεμάτων ήθιστε να παρίστατε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Καλώς ήρθατε κύριε Αρτουή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρίε και κύριοι, δεν πρόκειται να σας κάνω μια περιγραφή της κατάστασης. Είναι γνωστό ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη Και μάλιστα ήμουνα στη, την Πέμπτη στο Παρίσι και δεν περίμενα στο Παρίσι να ακούσω από Γάλλους μάλιστα Γεωργούς τόσα πολλά παράπονα στις αγορές που παρευρέθηκα Και τόση μεγάλη δυσαρέσκεια και δυσφορία για την παρούσα κατάσταση. Δεν το περίμενα αυτό. Η σημερινή συζήτηση και η συνεδρίαση μας είναι έκτακτη, γι' αυτό δεν θα χρονοτριβήσω άλλο. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Επίτροπο, μετά για δύο λεπτά στους συντονιστές και κατόπιν από ένα λεπτό στους συναδέλφους. Ελπίζω να δεχτείτε αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman, members. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα μαζί σας, αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής σας και ευχαριστώ που μου δίνει τη δυνατότητα να σας περιγράψω πώς έχουν εξελίξει όσον αφορά την κρίση στις αγροτικές αγορές. Το ζήτημα αυτό μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και από μόνο του δείχνει αυτό πόσο έχει κρατήσει η κρίση αυτή και πόσο βαθιά είναι. Προτού αναφερθώ σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατάστασης αυτής και πώς μπορούμε και πώς έχουμε μέχρι στιγμής ανταποκριθεί και πώς θα αποκριθούμε στο μέλλον, θα ήθελα να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις. Πρώτον, δέχομαι πραγματικά ότι η κρίση είναι πολύ έντονη, πολύ βαθιά και δέχομαι επίσης και τη δυσαρέσκεια των αγροτών μας. Ουδέποτε έθεσαν αμφιβόλο την σημασία και την, της κρίσης αυτής κύριε Μποβέ και πραγματικά δέχομαι ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε δει ότι η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη και δεχομένως να κρατήσει και περισσότερο καιρό από όσο προβλέψαμε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Συμβούλιο και θέλουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση για του αγρότε μα βάσει των ε, παραμέτρων που έχω θέσει στο παρελθόν και που θα, στις οποίες αναφερθώ λίγο ακόμα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ανισορροπίε στην αγορά όσον αφορά τον τομέα του χείριου κρέατο και τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιέσει υπάρχουν και σε άλλου τομεί, Πολύ δύσκολη κατάσταση για ορισμένα λαχανικά στην ε, Νότια Ευρώπη. Να σα πω λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι ε, υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να κάνω μια βαθιά ανάλυση της αγοράς, την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη για πάρα πολλά προϊόντα μας και δεν έχει ανακάμψει τόσο γρήγορα όσο ελπίζαμε ή όσο θα θέλαμε. Επομένω, δεν υπάρχει λόγο αυτή τη στιγμή να σα πω ότι όπω και σε άλλου τομεί οικονομία, έτσι και τομεί των αγροτικών προϊόντων, επηρεάζεται από μακροοικονομικέ ε, εξελίξει. Είναι χαμηλή η ζήτηση και αυτό με την σειρά του έχει ε, πολύ σημαντική επίπτωση στις τιμές. Ξέρετε ότι έχει μειωθεί πολύ σημαντικά η τιμή του πετρελαίου και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει ερνητικά τους ε, εμπορικούς μας εταίρους, όπως για παράδειγμα την Κίνα, η οποία έχει παρουσιάσει επιβράδυνση και θα επιβραδυνθεί ακόμα περισσότερο η οικονομία της και έχουμε επίσης και τις επιπτώσεις από το ρωσικό εμπάρκο που έχει αποκλείσει πάρα πολλά σημαντικά ευρωπαϊκά προϊόντα από τη ρωσική αγορά ιδίω για ορισμένες χώρες που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότερες εξαγωγές πήγαιναν προς τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει από πέρυσι να παρέμβει προκειμένου να υποστηρίξει τους αγρότες μου. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι τα μέτρα υποστήριξη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έγινε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το απόθεμα το οποίο υπάρχει για την κρίση, χρήματα τα οποία προορίζονται προς τους αγρότες, 90 εκατομμύρια ευρώ έχουν επιστραφεί προς τους αγρότες από το απόθεμα αυτό. Και μετά την εξέλιξη και την κλιμάκωση που είχαμε στον τομέα του γάλακτος και του χειρίου κρέατος, 500 εκατομμύρια ακόμα ευρώ χρησιμοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 420 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στοχευμένα στα κράτη-μέλη προ του προμηθευτέ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να βοηθήσουν του αγρότε. Ορισμένα από τα χρήματα αυτά δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί, επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πόροι οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί επαρκώ. 10 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή τη στιγμή μέτρα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτές τις στοχευμένες ε, χρηματοδοτήσεις. Πέρυσι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ε, να απομείναν πλεόνασμα από την προηγούμενη ε, περίοδο του προπολογισμού. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον αυτό το απόθεμα έχει χρησιμοποιηθεί και ενδεχομένω να πρέπει να χρησιμοποιηθεί το απόθεμα τη κρίση. Βλέπετε ότι τα χρήματα αυτά, όπω σα είπα, ανήκουν στου ίδιου του αγρότε και θα έχω καλέσει ήδη το Συμβούλιο και καλό και εσάς αυτή τη στιγμή να δούμε από κοινού πώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν περισσότερα μέτρα και αν θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το απόθυμα το οποίο προβλέπεται για την κρίση και ήδη σήμερα το πρωί ο πρόεδρο του Συμβουλίου ζήτησε από τα κράτη-μέλη να του πούνε αν πραγματικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το απόθεμα κρίση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα μέτρα και προκειμένου να προέλθουν περισσότερα κονδύλια από τον κοινοτικό προπολογισμό. Ήδη το Φεβρουάριο συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη για την κατάσταση στι αγροτικέ αγορέ και ζήτησα τότε από του υπουργού να προτείνουν οι ίδιοι νέα μέτρα τα οποία πιστεύουν ότι θα μπορούσαν από σήμερα να εφαρμοστούν. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει δράση μόνο όταν τις το ζητήσουν οι συνομοθέτες. Αν ε, αποφανθούν υπέρ το Συμβούλιο δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά να σεβαστούμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής, να δούμε ποιοι είναι οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί πόροι και να καταλήξουμε τελικά σε μια ευρύτερη συνένεση για τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτών. Η 25η Φεβρουαρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλουν προτάσει στα κράτη-μέλη. Και αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί πάνω από 100 ξεχωριστά μέτρα και η Προεδρία ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτά ως εξής. Επανεργοποίηση μέτρων που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν όπως ιδιωτική αποθεματοποίηση, χρησιμοποίηση, ανάκτηση κάποιων αποζημιώσεων, να χρησιμοποιηθούν παλαιότερες πρωτοβουλίες όπως πρακτικές κατά του αθέμητου ανταγωνισμού, προπαρασκευαστικές δράσεις όπως να, να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες παρακολούθησης ή νέα παρατηρητήρια και επίσης να έχουμε επίσης και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση παραγωγής, για παράδειγμα παραγωγής γάλακτος. Όσον αφορά τους διαφορετικούς τώρα που πλήττονται, συντοποιούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε κάποια διαρθρωτικά περισσότερα μακροπρόθεσμα προβλήματα και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κάποια πιο συγκυριακά προβλήματα. Οι υπηρεσίες μου αναλύουν τις προτάσεις που πέβαλαν οι Υπουργοί, που πέβαλαν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Πάντως ελπίζω ότι μέχρι το επόμενο Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο προκειμένου να βελτιώσουμε, τους, να βοηθήσουμε συγχωρείτε τους Ευρωπαίους αγρότες στη δύσκολη αυτή περίοδο. Προφανώ κάποιες ιδέες δεν είναι καινούριε. Επομένω, θα μπορούσα ήδη να απαντήσω σε κάποιες από τις ιδέες αυτές για παράδειγμα, να δημιουργηθεί μια εξαγωγική πίστοση προς τους γεωργούς προκειμένου να ευνοηθούν και να προωθηθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ήδη στα 14 κράτη-μέλη έχουμε τέτοια μέτρα, αλλά όχι ειδικά για τα γεωργικά προϊόντα, για τα αγροτικά προϊόντα. Θεωρώ ότι την πρόταση αυτή μπορούμε να την εξετάσουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο μέσο. Και ω προ αυτό, θεωρώ ότι ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας. Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη παρακολούθηση διαφόρων τομέων πέρα από το γαλακτοκομικό τομέα. Και αυτή την πρόταση την εξετάσω περισσότερο, διότι γνωρίζουμε ότι οι αγορέ αυτέ είναι αρκετά απρόβλεπτε και προφανώ θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί και οι αγρότε να έχουν αξιόπιστε πληροφορίε. Επομένως, ε, επίσης, η άλλη ιδέα η οποία υποβλήθηκε όσον αφορά την δράση των τρίτων κρατών, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, και πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και κάποια μέτρα προώθησης. Ήδη χρησιμοποιούμε ένα σημαντικό αριθμό από αυτών και ήδη έχουμε έναν έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρησιμοποιούνται για τον τομέα του χείριου κρέατος και για το γαλακτομικό τομέα. Επίσης, 250 εκατομμύρια ευρώ και 5 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια θα δοθούν στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί επίσης και η ζήτηση του γάλακτος, προϊόν, το οποίο συμβάλλει βέβαια και στη γενικότερη δημόσια υγεία και να ευχαριστήσω τον κύριο Τεραμπέλα για τη σχετική του έκθεση που συζητήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια άλλη πρόθεση επί τη οποία θέλω να αναφερθώ είναι η τιμή παρέμβαση, που πολλοί είπατε ότι θα πρέπει να αυξηθεί. Εγώ ήμουν πάντα συνεπής προς αυτό και δεν έχω αλλάξει ούτε πρόκειται να αλλάξω την άποψή μου. Εφαρμόζουμε την κοινή γεωργική πολιτική την οποία οι ίδιοι νομοθέτε επέλεξαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στι 12 Οκτωβρίου του 2011 είχαμε πει Είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουμε με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική για μια πιο βιώσιμη γεωργία. Επομένω, η αύξηση των τιμών παρέμβαση αποτελούν πολύ σημαντική αλλαγή στη ρότα που θα, ακολουθούσε, που θα έπρεπε να ακολουθήσει η κοινή γεωργική πολιτική. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όλοι δεχόμαστε ότι ο τομέας ο γαλακτοκομικό αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ανισορροπημένος. Επομένως λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση στην τιμή παρέμβασης, αλλά ακόμα και αν υπάρξει αύξηση στην τιμή ε, παρέμβασης, δεν θα πρέπει αυτό να επηρεάσει την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων συγκεκριμένων κρατών μελών. Αυτή η αύξηση τη τιμή παρέμβαση ενδεχομένως απλώς να προωθήσει συγκεκριμένα κράτη-μέλη και να αυξηθεί περισσότερο τελικά η παραγωγή των προϊόντων αυτών, των γαλακτομικών προϊόντων και να μην οδηγηθούμε στην ευκταία επιθυμητή μείωση τη παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο που ούτε πρόκειται να προωθήσω την πρόταση αυτή για αύξηση τη τιμή παρέμβαση. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λάβουμε κάποια άμεσα μέτρα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με κάποια μακροπρόθεσμα διαφορετικά μέτρα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια νέα task force υπό τον κύριο Βίρμαν, η οποία θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως η διαφάνεια της αγοράς, η πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδοτικά μέσα, καθώς επίσης και πρόσβαση στις προθεσμιακές αγορές, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στην διατροφική αλυσίδα ή ακόμα και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη κάθε φορά προσφεύγει στη δικαιοσύνη για διάφορα ζητήματα. Όλα αυτά τα ζητήματα ή τα περισσότερα από τα ζητήματα αυτά έχουν φυγεί ε, από τη δική σας Επιτροπή. Η Task Force Birman θα καταφέρει να προωθήσει περισσότερο τα ζητήματα αυτά και γι' αυτό το λόγο σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή την ομάδα εργασία, σε αυτή την Task Force και είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Βίρμαν θα χαρεί πάρα πολύ να συμμετέχει περισσότερα δική σα Επιτροπή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ξέρω ότι απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή σα είναι η δέσμη μέτρων για το γάλα που άρχισε να ισχύει από το 2012. Η αναθεώρηση προβλεπόταν για το 2018, αλλά ώψη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέα, θα πρέπει ήδη από το 2016 να γίνει αναθεώρηση τη δέσμη αυτή ε, για την παραγωγή γάλακτο. Η αναθεώρηση αυτή πιστεύω ότι ήδη από το φθινόπωρο του 2016 θα υποβληθεί στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε αν η δέσμη αυτή μέτρων για το γάλα θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από το 2020, προκειμένου να ευνοήσει κατά αυτόν τον τρόπο του παραγωγού. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα δεν έχουν πλήρω χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τι οργανώσει παραγωγών, προκειμένου να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών, των παραγωγών, στη διατροφική αλυσίδα. Ξέρω ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυ όλε τι εξελίξει αγροτικέ αγορέ και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η πρόοδος είναι πάρα πολύ μικρή. Ο ρυθμός της πρόοδου της διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ απογοητευτικός και με κάθε εβδομάδα που περνάει μειώνονται οι προοπτικές να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της θητείας του πρόεδρου Ομπάμα. Αυτό το οποίο λέω συνεχώς από τότε που έγινε επίτροπος ε, για τα ζητήματα αυτά, θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αν αυτή η συμφωνία επικεντρώνεται μόνο σε συγκεκριμένου τομεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια θετική συμφωνία και όχι μια κακή συμφωνία. Και σα διαβεβαιώ ότι οι πιο ευαίσθητοι τομεί δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να ανοιχθούν προ τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πρόκειται να προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση να ενισχύσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα προϊόντα τα οποία έχουν μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει συμφωνία με τι ΗΠΑ, συμφωνία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί και από τα 28 κράτη-μέλη και από τα μέλη προφανώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω, εσεί εναπόκειται σε εσά να αποφασίσετε τελικά τι θα γίνει. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και με άλλα κράτη-μέλη ιδίω όσον αφορά κάποια ευαίσθητα προϊόντα όπω η ζάχαρη, το βόλιο κρέα ή τα πουλερικά. Εγώ σε κάθε περίπτωση θέλω να προασπίσω τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικά βέβαια για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώ και οι διαπραγματεύσει αυτέ με τι χώρε Μερκοσούρ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδίω με του πιο ευαίσθητου τομεί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολύ δεινέ επιπτώσει στη γεωργία. Θεωρώ λοιπόν ότι και εδώ πάλι θα μπορούσατε εσεί να συμβάλλετε πολύ επικοδομητικά. Κύριε Πρόεδρε, πέρα από τα διεθνή τα ζητήματα θα πρέπει να θίξουμε και το ζήτημα τη Ρωσία και δεν έχουμε πρόσβαση πλέον στην αγορά τη Ρωσία. Όλοι γνωρίζετε για ποιου λόγου δεν ε, είναι δυνατή η πρόσβαση αυτή. Πάντω είναι βεβαιό ότι συνεχίζουμε τι προσπάθειέ μα προκειμένου να ξεκινήσουν οι εμπορικέ συναλλαγέ με τη Ρωσία. Συνεχίζονται οι επαφέ με τη χώρα αυτή και όπω είπε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Γιούγκερ έχει έρθει σε πολλέ περιστάσει σε επαφή με τον πρόεδρο Πούτιν προκειμένου να απελευθερωθεί το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Δυστυχώ όμω ελάχιστη πρόοδο έχει σημειωθεί. Στα πλαίσια λοιπόν της απαγόρευσης αυτής του εμπάρκο έχουμε προσπαθήσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείσουμε τη ρωσική πλευρά να αποδεχθεί τη δική μας την πρόταση, αλλά δυστυχώς οι προτάσεις αυτές, οι δικές μας προσφορέ προσφορές δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Συμφωνώ με την ησυχία σας, αλλά πάντως πρέπει να σας πω ότι το ότι δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να σημειώσουμε πρόοδο δεν οφείλεται σε εμά, δεν ευθυνόμαστε σε εμεί. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξομαλύνουμε τη σχέση μα με τη Ρωσία. Επίση, περιμένουμε ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα αποφανθεί τον Απρίλιο όσον αφορά το εμπάργκο τη Ρωσία για την υγειονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προφανώ είναι μια αιτίαση τη Ρωσία η οποία δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν βελτιώνεται, μολονότι αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε κάποια μέτρα, δεν πρόκειται να κάμψουν γρήγορα τιμέ των γεωργικών προϊόντων. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τι ανησυχίε των κρατών μελών και τι ανησυχίε των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στη βεβαιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να στηρίξει του Ευρωπαίου γεωργού και του Ευρωπαίου κοινοτρόφου. Όλα τα μέσα τα οποία παρέχουν σε μένα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δύο συνομοθέτες, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπω λοιπόν στις σημερινή συζήτηση προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι μελλοντικέ προοπτικές και ποια μέσα και ποια μέτρα θα μπορούσαμε να αναλάβουμε για το μέλλον. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πρέπει να σας πω όμως ότι τα μέσα αυτά τα εργαλεία είναι περιορισμένα. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που έχουμε και πώς θα καταφέρουμε να καλύψουμε χρηματοδοτικά και όλες οι υπόλοιπες προκλήσεις που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν μας δίδεται η κατάλληλη ευκαιρία να ακούσουμε ποια μέτρα εσείς ως μέλη της Επιτροπής αυτής θα μπορούσατε να προτείνετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιληθεί η φυστάμενη κρίση. Προσβλέπω λοιπόν στην παρουσίαση των μέτρων αυτών, αλλά σας παρακαλώ πολύ στην παρουσίασή σας λάβετε υπόψη και τις παραμέτρους και τις προποθέσει που έθεσα παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Όπω σα είπα, έχουμε 8 συντονιστέ από 2 λεπτά καθένα, 16 λεπτά και μετά έχουμε 9 ομιλητέ από 1 λεπτό, θα φτάσουμε στα 45 λεπτά, να αφήσουμε 10-15 λεπτά για τι απαντήσει ε, του Επιτρόπου. Δεν θέλουμε να παρατείνουμε το χρόνο της ε, συνεδρίασης. Άρα το τελευταίο τέταρτο θα πρέπει οπωσδήποτε να το αφήσουμε στον Επίτροπο για να μπορέσει να απαντήσει. Ο κύριος Αλμπερντές, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι δύσκολο μέσα σε δύο λεπτά να παρουσιάσουμε όλοι μας την επιχειρηματολογία Σα ευχαριστούμε για όσα μα είπατε σε σχέση με την κρίση και θα ήθελα να λάβω κι εγώ ε, θέση του θέματος. Αναφέρω την προσωπική μου θέση για τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Το τωρινό σύστημα ε, παρεμβάσεων ε, θεωρώ ότι είναι σφαλμένο. Θα προτιμούσα να καταργηθεί η τιμή παρέμβαση για το γάλα. Θα θέλαμε να έχουμε ένα ad hoc σύστημα και κατά περίπτωση να ε, ε, αποφασίζετε αν το γάλα πρέπει να αποσύρεται από την αγορά. Το εμπόριο μπορεί να αποφασίζει ε, αν χρειάζεται παρέμβαση. Νομίζω ότι επί αυτή τη πρέπει να αποφασίσουμε ποιο σύστημα λειτουργεί καλύτερα. Επίσης, για την τιμή του βουτύρου πριν από τέσσερα χρόνια ήταν στα τέσσερα ευρώ. Έχει ανέβει όμως ε, η τιμή και έχουμε υποκατάσταση προϊόντων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με τι τιμή μπορεί να γίνει η μεταποίηση ε, των προϊόντων, τόσο ώστε να μην έχουμε υποκατάσταση ευρωπαϊκών προϊόντων από προϊόντα τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα Juncker και να δούμε ε, πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, παραγωγής και επεξεργασίας ε, γάλακτος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την μεταποίηση και να τις εξασφαλίσουμε σε σχέση με τους κινδύνους εξαγωγών. Ε, το επίπεδο των δασμών επίσης είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί και δεν μπορούμε να ε, υποχωρήσουμε έναντι των Αμερικανών στα θέματα των δασμών. οι Αμερικανοί μαζί με τους Ρώσους ε, ε, συνεργάζονται σε προγράμματα για το διάστημα χωρίς να μποϊκοτάρουν τους Ρώσους. Δεν μπορεί να μποϊκοτάρουν εμάς λοιπόν και μας υποχρεώνουν ε, να εφαρμόζουμε εμείς μποϊκότ έναντι των Ρώσων για θέματα όπου θα μας συνέφερε να συνεργαζόμαστε με τους Ρώσους. Ξέρω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεκάστρο. Παρακαλώ. Βλέπετε πίσω τα χρονόμετρα. Παρακαλώ μην περιβείτε το χρόνο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ ο Επίτροπος, ο οποίος παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια κρίση, μια βαθιά κρίση. Η Επιτροπή μας όμως σας το έχει πει εδώ και αρκετό καιρό κύριε Επίτροπε και ήδη είχαμε εκφράσει στο παρελθόν τις ανησυχίες μας σε σχέση με την δεινή αυτή κατάσταση. Ξέρετε ότι ο τομέας του χείριου κρέατος, ο τομέας του γάλακτος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση που παρόμοιά της δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ καταρχάς που παραδέχεστε την σοβαρότητα της κατάστασης κύριε Επίτροπε. Πρέπει όμως να δούμε, όπως το είπατε κι εσείς, ποιους κανόνες έχουμε στη διάθεσή μας και πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, απέναντι στην πληθυκότητα αυτή των αγορών, νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση για τη διαχείριση του κινδύνου. Και δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση αν αυτή δεν γίνει υπό το φως ε, μιας ενδιάμεσης αναθεώρησης της πολιτικής που ακολουθούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η κοινή ορική πολιτική έχει κάποια εργαλεία τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις όπου μειώνονται, κατακριμνίζονται μάλιστα οι τιμές των προϊόντων και δεν καταφέρουν να αποκριθούν οι αγρότες μας. Και όπως το έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και στα πλαίσια της ίδιας της αναθεώρησης κοινή γεωργικής πολιτικής, Ορισμένες ε, χώρες του Συμβουλίου δεν κατάφεραν να αποδεχθούν τις δικές μας τις προτάσεις ή την πρόταση του κυρίου Νταντέν όταν είχαμε πει τότε στο παρελθόν ότι θα έπρεπε να είχαμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την πτυτικότητα και την ε, διακύμαση αυτή των τιμών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια λύση αυτή τη στιγμή και προφανώς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε στις ποσοστώσεις γάλακτος, να παίξουμε δηλαδή με την προσφορά των προϊόντων. Ξέρετε ότι ε, οι ποσοστώσεις γάλακτος που ίσχυαν στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ίσχυαν ισότιμα για όλες τις χώρες. Το τίμα όμως όλες οι χώρες το καταβάλουν τώρα. Επίσης δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή τη στιγμή μια τόσο χαμηλή τιμή στον παραγωγό τη στιγμή που δεν έχει ισότιμα μειωθεί και η τιμή για τον καταναλωτή. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι οι αθέμητες πρακτικές στα πλαίσια της διατροφικής αλυσίδας και ελπίζω ότι με την πρόταση της κυρίας Μαγκίνες θα καταφέρουμε να έχουμε συγκεκριμένε προτάσεις και δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να δραστηριοποιηθούμε και να αρχίσουμε να έχουμε επιτάπητο συγκεκριμένε πλέον προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Και καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχετε ήδη λάβει το σχόλιο των κρατών μελών επί των προτάσεων θα δεξάσετε την επόμενη εβδομάδα. Ε, Πώς σας φαίνονται οι απαντήσεις που λάβατε, υπάρχουν καινοτομίε αυτές, ε, ε, σας υπέβαλα καμία φαϊνή ιδέα που δεν μπορέσαμε εμείς να σκεφτούμε. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική αποθεματοποίηση, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο. Θα έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο μέχρι τον Απρίλιο. Υπάρχει πρόταση για την παράταση τη ιδιωτική αποθεματοποίηση. Γιατί αν περάσουμε σε σύστημα πληστηριασμών θα γίνει μια μειοδοτική ε, προσπάθεια, ένας σημειοδοτικό ανταγωνισμός, ε, να τα ρίξουμε προς τα κάτω, κάτι που θέλει είναι βάρος των γαλακτοπαραγωγών. Και διαφωνώ σε ό,τι αφορά την παρέμβαση μαζί σα, Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, είναι πολύ παλιά αυτή η αντιπαράθεσή μας. Νομίζω ότι ένα από τους τομεί όπου μπορούν ε, οι γεωργοί να ελπίζουν σε αύξηση των τιμών είναι το θέμα κατάσταση στα λοιπάσματα. Γιατί όταν είχαμε υψηλές τιμές πετρελαϊκών προϊόντων, είχαμε πει ότι ακριβώς επειδή τα λοιπάσματα περίχαν και πετρελαϊκά προϊόντα, γι' αυτό ήταν τόσο οι τιμέ τους. Τώρα, ένας εκπρόσωπος από τη λοιπασματοβιομηχανία ε, είπε ότι οι τιμές των λοιπασμάτων προσαρμόζονται στην αγορά και την, ε, στην προσφορά και τη ζήτηση και έχει μειωθεί. Κανονικά θα πρέπει μάλλον να έχει μειωθεί, γιατί έχει μειωθεί και η ε, το ύψος των πετρελαϊκών προϊόντων. Μήπως λοιπόν θα, μπορέσουμε να, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στον τομέα αυτό, σε ό,τι αφορά το χείριο κρέας. Λυπάμαι γιατί δεν καταφέραμε να το συμπεριλάβουμε ε, στην ε, εγκαίρω στην ημερήσια διάταξη. Θα μπει στις 3 το απόγευμα την Πέμπτη, θα αναποσιάζετε και εσείς και πάρα πολύ. Ε, συνάδελφοι, ενώ η κατάσταση για το χείρο κρέας και η χειροτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και ελπίζω να γίνει κάτι το συντομότερο δυνατό, γιατί πραγματικά είναι τρομερό το πρόβλημα στο χείριο κρέας. Επίσης, ε, ε, μία τράπεζα από την εκλογική μου περιφέρεια είχε στείλει επιστολές σε γεωργούς που βρίσκονται σε την κατάσταση. Και φαίνεται ότι έχουμε πιάσει πάτο στην κατάσταση αυτή Μερικοί ε, αγρότες βρίσκονται με το μαχαίρι στο λαιμό και δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρότατα προβλήματα και κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα υπάρχοντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, ζητούν να επιδοτηθούν τιμές παραγωγή και αυτό μας οδηγεί βήματα προς το παρελθόν και δεν βοηθά τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά και δεν θέλει να δώσει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση πάνω από τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουν ε, δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρχές του 2015. Η μόνη διαρθρωτική λύση είναι να γίνει πιο ανταγωνιστικός ο τομέας της διοργίας στην παγκόσμια αγορά. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε πολλούς τομείς. Καταρχήν, και το πιο σημαντικό ίσως, είναι οι καλύτερες νομοθετικές διατάξεις. Χρειαζόμαστε απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε και άλλους νόμους που θα είναι προσανατολισμένοι προς τους στόχους που επιθυμούμε. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη νομοθεσία για να εξοικονομήσουμε κόστος, κόστος λιπασμάτων παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώντα περισσότερο ζωική, ζωική κοπριά. Επίσης είναι σημαντικό οι αγρότες ε, να κάνουν επενδύσεις για να ανταποκρίνονται ε, ε, στις απαιτήσει της αγοράς. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν κατά νου και τη δική τους εθνική νομοθεσία για να εφαρμόζουν και εκεί την καλύτερη νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη πολύ συχνά μόνο περισσότερα χρήματα ζητούν από τις Βρυξέλλες και δεν δίνουν επικοδομητικές λύσεις. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε νέες αγορές και να συνάψουμε σωστέ εμπορικέ συμφωνίε, το συντομότερο δυνατόν. Τρίτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών στην, αλυσίδα, στην τροφική αλυσίδα και το αποτέλεσμα της Task Force για τις γεωργικέ αγορέ είναι πολύ θετικό και είναι πολύ ενδιαφέρον και ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό να οργανωθούμε καλύτερα, να οργανωθούν, καλύτερα οι συνεταιρισμοί των αγροτών. Οι παραγωγοί μπορούν να πολλούν περισσότερο άμεσα τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς πολλούς ε, ενδιάμεσους. Και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και περισσότερο καινοτόμοι. Ευχαριστώ. Κυρία Σένρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο στην πραγματικότητα. Γιατί είπε, είπε ότι πήγε στην Γαλλία και διαπίστωσε την κακή κατάσταση που υπήρχε. Γιατί ποτέ, κύριε Πρόεδρε, είπατε και εσείς ότι δεν ακούσατε τόσα παράπονα από Γιώργους. Ίσως γιατί δεν μας ακούει ο Επίτροπος που συχνά λαμβάνουμε το λόγο και επισημαίνουμε την κατάσταση συνεδριάσης τη ε, θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και τον Επιτροπο Χόγκαν στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματικότητα, γιατί επιτέλου αναγνώρισε ότι διανύουμε κρίση και μάλιστα βαθύτατη κρίση. Μέχρι πρόσφατα μάλιστα φαίνεται ότι δεν παραδεχόταν αυτή την κατάσταση της κρίσης ο Επίτροπος. Και με εκπλήσει το γεγονός ότι και ο Επίτροπος Χόγκαν αλλά και οι προλαλήσαντες δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε μία από τις βασικές συνέπειες ή σε μία από τις βασικές, θα μέσα τους βασικούς λόγους της κατάστασης, ε, που είναι η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή φταίει σε μια απο τις βασικες θα μεσα στους βασικους λογους της καταστασης που ειναι βαθμό για τη σημερινή κατάσταση. Και βλέπουμε ότι έχουμε μία από τα ίδια. Έχουμε τις ίδιες λύσεις ε, με αυτές που είχαμε πριν από τρία χρόνια, από ένα χρόνια, από έξι μήνες, από δύο μήνες. Όλα για τα ίδια μιλάμε, όλο τα ίδια προτείνουμε και τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Γιατί λοιπόν δεν παραδέχεστε το λάθος που κάνατε με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, γιατί δεν διερευνάτε και άλλες λύσεις σαν αυτές που προτείνουν οι γεωργοί, οι γεωργικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μερικοί ευρωβουλευτές. Πρόκειται για νέες ε, λύσεις για αξιοποίηση της ρύθμισης της παραγωγής και της ρύθμισης των αγορών. Γιατί αν συνεχίσουμε με τις ε, προτινόμενες λύσεις είναι ε, σαν να κατασπαταλούμε το, τα δημόσια κονδύλια, σαν να κοροϊδεύουμε και να παραπλανούμε το τομέα και να προτείνουμε ψευδολύσεις ενώ ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η ταχύτατη εξαφάνιση και η οικονομική εξολόθρευση ε, εκατοντάδων γεωργών και των οικογενειών τους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη συζήτηση που είχαμε για το γαλακτοκοπικό τομέα μετά από μία επίσκεψη που είχε κάνει η Γεωργική Επιτροπή. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπατε και εσεί, υπάρχει μια κρίση και άλλοι συνάδελφοι συμφωνούν. Πριν από λίγε εβδομάδε είπατε ότι υπάρχουν στρεβλώσει τη αγορά και μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών. Ίσως είναι η μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και δεν υπάρχει και φως στην άκρη του τούνελ. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Δυστυχώς σήμερα το βράδυ δεν άκουσα καμία λύση από εσά. Είπατε ότι μπορούμε να σκεφτούμε να επαναφέρουμε τις εξαγωγικές πιστώσεις. Είναι σαν να γυρνάμε στη δεκαετία του 70, της περασμένης χιλιετίας. Βουνά από βούτυρο, λίμνες από γάλα κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορούν οι φορολογούμενοι απάπειρον ε, να δίνουν χρήματα. Δεν έχουμε κρίση της ζήτησης, αλλά έχουμε υπερπροσφορά. Αυτό δημιουργεί την κρίση. Ε, υπευλήθησαν και προτάσεις στο Συμβούλιο από τη γαλλική πλευρά για να... Ε, προσπάθεια ε, ρύθμιση, ρύθμισης της αγοράς. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε στις τεράστιες ποσότητες. Πρέπει να δούμε και ποια είναι η πιο φτηνή λύση. Να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε και από πολιτικής πλευράς. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Η ποιότητα είναι αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε στην Ευρώπη. Με την ποιότητα θέλουμε να προσεγγίσουμε τον ε, καταναλωτή στην Ευρώπη. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ε, ότι ε, εν μέρει είναι ψέμα ότι το εμπάργο της Ρωσίας είναι η αιτία όλων των προβλημάτων. Δεν μπορούμε να λέμε στους αγρότες ότι αν αρθεί το εμπάργο ξαφνικά θα γίνουν όλα καλύτερα. Νομίζω ότι θα πρέπει προς τους αγρότες να είμαστε ειλικρινείς και να δείξουμε ποιες είναι οι σωστές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Εγώ αντίθετα με τους άλλους δεν θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Γιατί οι, οι Ευρωπαίοι Γεωργοί, κυρίως οι Γάλλοι, περνούνταν πάντα εξαιτία σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται, κύριε Επιτρόπε, ξεκίνησε μία έρευνα για, τον όμιλο Intermarché για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το μόνο της έγκλημα ήταν ότι έκανε μία χειρονομία Προ του Ευρωπαίους, προς τους Γάλλους γεωργίους και κτηνοτρόφους και προσπάθησε να στηρίξει το χείριο τομέα που εσεί ε, και οι μέτεροι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρατε σε δύσκολη θέση. Το μόνο του έγκλημα ήταν ένα οικονομικό πατριωτισμό ε, βοηθώντα του ε, Γάλλου χειροτρόφου. Σταματήστε επιτέλους κύριε Επιτροπή, σταματήστε αυτή την έρευνα που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βοηθήστε του Γάλλου διανομή και γεωργού γιατί η κατάσταση είναι τραγική για όλο και περισσότερους επαγγελματίες και βέβαια ε, κατηγορούμε συνήθως ε, τα, ε, τους μεγάλες, μεγάλες αλυσίδες ενομής, αλλά μερικοί όπως η Ιντερμασί δείχνουν ευαισθησίες και πολλοί πιστεύουν ότι ε, η ΚΑΠ δεν εξασφαλίζει δίκες τιμές των γεωρικών προϊόντων. Θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική, αλλά να μην καταπνίξουμε την παραδοσιακή γεωργία. Οι στόχοι της ε, πολιτικής, όπως προβλέπει η έκθεση Μάσχολτ, ε, ουσιαστικά περιορίζονται στην αποδοτικότητα και στην παραγωγικότητα. Οπότε ο ΕΚΙΑ λίμωνο για τους παραγωγούς και τους χωρικούς. Επίσης έχουμε και το ΤΤΙ που επίσης απειλεί σοβαρά την ε, Γαλλική Γεωργία. Και μάλιστα όλοι οι εμπειρογνώμονες, ακόμη και οι Αμερικανοί, συμφωνούν ότι θα γονατίσει η συμφωνία αυτή τους γεωργούς μας. Η υπογραφή του TTIP θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μια ανικανότητα και στη χειρότερη μια προδοσία εις βάρος των Ευρωπαίων Γεωργών. Πριν από ε, λίγε εβδομάδε είπατε σε μια ερώτησή μου ότι δεν θα πρέπει οι Γάλλοι Γεωργοί να παραπονούνται για την κατάσταση. Κι όμως ε, η πραγματικότητα σας διαψεύδει, κάνατε λάθος. Θα ακούσετε επιτέλου ε, την φωνή της απελπισίας των Γεωργών και θα προσπαθήσετε επιτέλους να δείξετε την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ολοκληρώσαμε τους, ε, με τους συντονιστές. Ο κύριος Σάντος για ένα λεπτό όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Ε, ευχαριστούμε για την προθυμία σας ε, να έρθετε για ανταλλαγή απόψεων. Ε, πρόκειται για μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί από την αρχή τη κοινοβουλευτική θητεία και έχουν σχεδόν στραγγαλιστεί γαλακτοπαραγωγή. Είναι, πουλάν ε, σε τιμή κάτω του κόστους και μάλιστα τώρα θα πρέπει να εξαναγκάζονται να μειώσουν ε, την προσφορά για να εξισορροπήσουν τις τιμές. βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και απειλείται ο γεωργικός ιστός, η εκτινοτροφικός ιστός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με πλήγμα φοβερών προϊόν, σημαντικών προϊόντων όπως ε, του γάλακτος, του τυριού, του βουτύρου, θα πρέπει να βρούμε μια συνολική λύση για να εξασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό του κλάδου. Έχουμε πλεόνασμα παραγωγής, αλλά ε, δεν φταίνε για όλη η γεωργία γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε τα μέτρα που ελήφθησαν, γιατί στην αλυσίδα των αξιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος της παραγωγής, αλλά και το κόστος της διανομής. Κύριε Επίτροπε, συγκεκριμένα τι μέτρα πρόκειται να λάβετε για να βοηθήσετε άμεσα τους παραγωγούς γάλακτος. Ευχαριστώ. Κύριε Μίλλορ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποια θέματα. Πολύ συχνά στη Γερμανία τονίζεται ότι δεν χρησιμοποιείται η υπάρχουσα ε, ρευστότητα, αλλά χρησιμοποιείται ο κανόνας ε, de minimis. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, ποια είναι η γνώμη σας για θέματα εξασφάλισης των επιχειρήσεων και για το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Dairy Matching. Πώς μπορούμε εμείς ε, να υποστηρίξουμε τους Ευρωπαίους αγρότες. Το επόμενο ερώτημα επίσης είναι πολύ ε, σημαντικό. Ε, θα, παρεμβεί, θα παρεμβείτε στο ρυθμιστικό επίπεδο για το λιανικό εμπόριο των ειδών διατροφής. για τις λιπαρές ουσίες ε, θα κάνετε παρέμβαση για να υποστηρίξετε την βιομηχανία μεταποίησης. Ήδη ο Άλμπερτ Ντες ανέφερε αυτό το θέμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος ici θα ήθελα να αναφερθώ στις πραγματικές δυσκολίες που επιτόπου αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Αυτή τη στιγμή δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση σε εικασίες που έχουν να κάνουν με τη μεταβλητότητα των τιμών. Αναφέρομαι σε άντρες και γυναίκες που υποφέρουν σε καθημερινή βάση, δεν καταφέρουν χρηματικά να τα βγάλουν πέρα και επίση βλέπουν ότι δεν υπάρχουν προοπτικές αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή η ίδια αγορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί από μόνη της. Ξέρετε ότι ε, υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις που ήρθαν στη δική μου την ε, ε, περιφέρεια, άφησαν μπροστά από το γραφείο μου δύο χείρους. Τι μπορώ να πω στους ανθρώπους αυτούς, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι κανόνες οι οποίοι στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Τι μπορώ να προτείνω ως Ευρωβουλευτής σαν λύση στους ανθρώπους αυτούς. Δυστυχώ, πώς μπορώ να του πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του γυρίζει την, πλάτη και ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αρνείται τελικά στου ανθρώπους αυτούς να μπορούν να δουλέψουν τη γη τους, να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις γεωργικές αγορέ. Κύριε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που μας έκανε μια σαφή παρουσίαση. Βέβαια δεν μας είπε όλα όσα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά τουλάχιστον ήταν σαφής. Η ερώτησή μου είναι απλούστατη. Δεδομένου ότι οι γεωργοί ε, παράγουν για να πουλούν και υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη ε, αναζήτησης και διέξοδο διεθνώς ε, των προϊόντων τους, τι πρόοδος έχει γίνει σε ό,τι αφορά την ανέβρεση νέων αγορών για την διάθεση των προϊόντων και μάλιστα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ κύριε Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Για το θέμα των εξαγωγικών πιστώσεων που αναφέρατε, θα ήθελα να ακούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί ήδη είχαμε μια τέτοια λύση και σε πολλές περιπτώσει δεν ήταν ε, το μέσο το οποίο χρειαζόμασταν. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να κατακλειστούν αγορές από ευρωπαϊκά προϊόντα ε, τη στιγμή που αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τις χώρες ε, του τρίτου κόσμου που πεινάνε. οι αλυσίδε ενδεχομένω είναι η καρδιά του προβλήματο. Το 80% τη παραγωγή στην Αυστρία κυκλοφορεί και διακινείται μέσω τριών μεγάλων αλυσίδων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και το τι πραγματικά χρειάζονται οι αγρότες. Θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση για το θέμα της Ρωσίας, το οποίο επίσης αναφέρατε. Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν και πάλι οι αγορές. Ποια είναι η εκτίμησή σας. Τι χρονικό ορίζοντα βάζετε. Ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Επιτροπέ να σας επισημάνω ένα πρόβλημα που αφορά περισσότερο τον Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Προϊόντων. Αφορά τις πατατοπαραγωγούς. Πριν από 15 χρόνια είχαμε την τρίτη θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ε, παραγωγή ε, τροφίμων. Μετά τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις και εξαιτία ενό παρασίτου πατάτε, είμαστε η μόνη χώρα που προσχώρησε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποχρεωμένη να δεχθεί ειδικέ εργαστηριακές ε, έρευνε προκειμένου να διαθέσει τα προϊόντα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι προποθέσει. Είμαστε η μόνη χώρα που υφιστάμεθα τέτοιε προποθέσει και μάλιστα έχει μειωθεί πέντε φορές η παραγωγή παρόλο που η βακτηριακή κατάσταση των προϊόντων μα είναι παρόμοια με αυτή των άλλων χωρών. Ε, η Πολωνοί παραγωγοί βρίσκονται σε δυσμενή θέση, υφίστανται αρνητική διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει επιτέλου να σταματήσουν αυτέ τι διακρίσει ει βάρο των Πολωνών παραγωγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που συζητάτε αυτά τα προβλήματα μαζί μα Θα ήθελα να προσθέσω κάποια θέματα σε αυτά τα οποία έχουν ήδη ακουστεί. Όσον αφορά τα εθνικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν, πρόσθετα εθνικά μέτρα. Αν ένα κράτος μέλος ε, θέλει να δώσει ε, κάποιες διευκολύνσεις στους αγρότες. Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στα κάτι μέλη να λάβουν κάποια μέτρα υπέρ των αγροτών. Όταν μιλάτε ε, για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Ε, θα μπορούσα να το υποστηρίξω αν ε, εννοείται εξαγωγικές εγγυήσεις για την παρέμβαση δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε θέματα πληστηριασμών για ποσότητες γάλακτος θα μπορούσαν να δοθούν στους πρόσφυγες, παραδείγματος χάρη. Και μια τελευταία ερώτηση για τις ε, ε, εμπορικές αλυσίδες. Ε, υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες όπως το Aldi στη Γερμανία και πολύ συχνά υπάρχουν και θέματα dumping που πρέπει να λυθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω κύριε Επίτροπε αν μας ακούν σήμερα οι Γεωργοί. Αλλά έχω την αισθησία ότι εσείς τουλάχιστον κοφεύετε. Γιατί ήμουν στην έκθεση Γεωργίας ε, την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία και όταν μου λέτε μην περιμένετε από μένα να αυξηθεί η τιμή ε, παρέμβασης δεν ήταν αυτό που άκουσα στις τρίμερες ε, συναντήσεις που είχαμε επαγγελματίε και γεωργούς. Θα πρέπει να δράσουμε και μάλιστα πάρα αυτά ε, κραυγάζουν οι γεωργοί και όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της 14 Μαρτίου θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνε σας κύριε Επίτροπε. Έχετε τα εργαλεία στη διάθεσή σας και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Δεν θα πρέπει να περιμένετε να σχηματιστεί πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να τα χρησιμοποιήσετε. Ξέρετε ότι θα πρέπει να επέμβετε στις κοινέ οργανώσεις αγοράς και στον όγκο των προϊόντων θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε το άρθρο 221 και το άρθρο 222. Έχετε αυτά τα εργαλεία να τα αξιοποιήσετε ώστε κατεπηγόντως να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του Γεωργό και στην κρίσιμη κατάσταση που διανύουμε όλοι σήμερα από κοινού. Ευχαριστώ. κυρία Γιλέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που άκουσα σήμερα ότι εστερνίζεστε και εσείς την άποψή μας ότι η γεωργία διανύει κρίση. Είναι σημαντικό και έστω και αυτό είναι πρόοδος, ότι συμφωνούμε ότι υπάρχει κρίση, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να την αντιμετωπίσουμε. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να ανασκομποθούμε και να ξεκινήσουμε μια σοβαρή μεταρρύθμιση των μηχανισμών που έχουμε για την αγορά των απορροκυπευτικών. Και η μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στο επιτελείο σας με το ε, εκτελεστικό κανονισμό 1543 του 2011 δεν νομίζω ότι είναι ε, η σωστή λύση, ούτε αυτό ζητάνε οι διάφοροι τομείς. Το είπαμε και στον εκπρόσωπο τη Επιτροπή στην προηγούμενη μα συνεδρίαση. Δεν είναι σωστή αυτή η λύση. Δεν πήρε το σωστό δρόμο η μεταρρύθμιση του κανονισμού 543 του 2011, του εκτελεστικού κανονισμού. Θα πρέπει να παταχθούν οι αθέμητες πρακτικές των αλυσίδων διανομής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού, είναι δύσκολο το θέμα, δυσεπίλητο, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Επίσης, η αστάθεια των τιμών, οι τρομερές και τι γίνεται με την επιστημιστική αλυσίδα σήμερα. Επίσης, μία τελευταία ερώτηση προς τον Επίτροπο. Όπως είπε ο κύριος Νίκολσον, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να έχουμε μια συζήτηση ε, για το χείριο ε, κρέας, για, το, για τη χειροτροφία, πέμπτη απόγευμα στις 3, όταν θα είμαστε 3 και ο Κούκος. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να δείξουμε ότι δείχνουμε σεβασμό προς τα αιτήματα των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, γιατί δεν είναι σωστή αυτή η λύση που βρέθηκε. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μα είπατε, μα ζητήσατε μάλλον να σα ανακοινώσουμε κάποια θετικά μέτρα, αλλά από εσά το μόνο το οποίο άκουσα είναι να αναδημιουργηθούν νέε εξαγωγικέ πιστώσει, κακή ιδέα κατά την άποψή μου, για τον πολύ απλό λόγο γιατί στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη αυτή πολιτική δεν επιτρέψαμε σε κάποιους μικρούς Αφρικανούς γεωργούς να καταφέρουν να αναπτυχθούν, να καταφέρουν να είναι αυτόνομοι και να μπορούν να ανταγωνιστούν τα δικά μας προϊόντα. Επομένω δεν υπάρχει λόγος να επανέλθουμε στο μέτρο αυτό. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, εγκαταλείπουμε του ε, ρυθμιστικού μηχανισμού, ποσοστό για το γάλα για παράδειγμα, ποσοστό για τη ζάχαρη του χρόνου και παράλληλα όμω ανοίγουμε χωρί καμία προστασία την αγορά μα. Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Πίτροπε δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντική η δική μα ε, η δραστηριότητα, εφόσον από ό,τι φαίνεται στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είμαστε το τελευταίο διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έχουμε στρατηγική μεταρρύθμιση για τα επόμενα 20 και 30 χρόνια τη κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να έχουμε μια γεωργία σε ανθρώπινη κλίμακα η οποία να είναι βιώσιμη. Κύριε Επίτροπε, για πολλά πράγματα θα ήθελα να σας μιλήσω, για τη ρύθμιση, τις νομαστικές ρυθμίσεις, για τις τιμές, αλλά αυτό το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε είναι 600 αγρότες που αυτοκτόνησαν στη Γαλλία μέσα σε αυτή τη χρονιά. 600 αυτοκτονίες. Σχεδόν όσα και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Δεν έχω χρόνο, μόνο 40 δευτερόλεπτα. Ας αφιερώσουμε λοιπόν ένα λεπτό σιωπής στα θύματα αυτά, 600 αγρότες που αυτοκτόνησαν. ενό λεπτού σιγή. Je Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο Κύριε Επίτροπε, όπω όλοι γνωρίζουμε και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στη Γεωργία. Και εσεί αναζητείτε λύσει και εγώ αναζητώ λύσει και η Επιτροπή μα αναζητεί λύσει. Πήγα για ψώνια λοιπόν και αγόρασα λύσει. Τσάι αγόρασα, από την Ινδία, μπανάνες από την Καραϊβική, σοκολάτα από τη Γάνα, καφέ από την Κένια. Αυτά είναι τα ψώνια μου. Αυτό το οποίο έχουν από κοινού είναι το σήμα του δίκαιου εμπορίου, fair trade. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι μια εγγύηση ότι είχαν σωστή τιμή οι αγρότες για αυτά τα προϊόντα. Τι άλλο ψώνισα. Λουκάνικα από την Πολωνία, μήλα από την Ιταλία, τυρί από την Αγγλία και γάλα από τη Γαλλία. Και δεν έχω εγγύηση ότι για αυτά τα προϊόντα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί είχαν δίκαιη τιμή και μάλιστα μπορεί να ήταν και χαμηλότερη τιμή από το κόστος παραγωγής τους. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν για την Επιτροπή μας και για τι ενώσει των αγροτών και για, τον, για τους αγρότες τους ίδιους. Πριν από 15-20 χρόνια, λίγες μη κυβερνητικέ οργανώσεις κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το σήμα χωρίς ε, χρήματα από το δημόσιο κορβανά και κατάφεραν να επιτύχουν να υπάρχει εγγύηση για μια δίκαιη τιμή στους αγρότες στον αναπτυσσόμενο κόσμο ενώ εμείς με όλες μας τις ικανότητες και την επιρροή μας και τα χρήματά μας δεν έχουμε καταφέρει να δίνουμε δίκαιη τιμή στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ακριβώς εκεί βρίσκεται η απάντηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα σήμα δίκαιου εμπορίου και δίκαιας τιμής για τους παραγωγούς στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μας ευνηδιάσατε. Μας ευνηδιάσατε τόσο πολύ που δεν κατάφερα να μετρήσω και το χρόνο σας. Η κυρία Ντότζ. Σας ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και σας ευχαριστώ για την προθυμία σας ε, να αναζητήσετε λύσεις. Δύο ερωτήσεις. Θα υποβάλλετε πρόταση για την προσωρινή αύξηση του, της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποπληρωμένο γάλα σε σκόνη. Και αν περάσουμε στη διαδικασία πληστηριασμού, με τι μέτρα θα φροντίσετε να αποτρέψετε μείωση της συνολική τιμής του γάλακτος. Πολλά κρατημέλη εφαρμόζουν εσκεμμένως ε, την αύξηση της παραγωγής γάλακτος. Στη Βόρεια Ιρλανδία όμω, κάποιοι ε, γεωργοί αυξάνουν την παραγωγή, όχι επειδή έχει βελτιωθεί η αγορά, αλλά σε μία απόπειρα να έχουν περισσότερα ρευστά. Ε, η γεωργοί όμως που έκαναν επενδύσεις ε, και υφίστανται μακροχρόνια ζημίες, ελάχιστες ελπίδες έχουν για βιώσιμο μέλλον όταν ε, υπερχρεώνονται. Πώς μπορεί να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους τους ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν με κάποια ελαστικότητα την παρούσα κρίση και να ταινίσουν το μέλλον τους. Η κυρία Ριμπέιρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τιμές που είχαμε σε περιφερειακές χώρες, κυρίως στις Αζόρες. Μειώνονται συνεχώς οι τιμές, ιδιαίτερα στο γάλα, και δεν έχουμε καμία, κανένα αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Υπάρχει μια διακοπή γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία. Θα πρέπει να ξαναρχίσω. Ναι. Κύριε Επίτροπε, έχουν καταρρεύσει οι τιμές προϊόντων στις περιφερειακές χώρες, κυρίως στην Πορτογαλία και δι στις Αζόρες. Ε, μειώνονται συνέχεια οι τιμές του παραγωγού. Και μάλιστα έχουμε όλο και μεγαλύτερο έλεγχο τη παραγωγή. Κάτι που αν δεν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει κανένα αντίκτυπο. Και ουσιαστικά θα πληγούν ε, μόνο γεωργοί εκείνοι που μειώνουν την παραγωγή, ενώ άλλοι θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη δική του παραγωγή δημιουργώντα ανταγωνιστικό πλονέκτημα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, τις να μειώσουν την ε, την εξάρτησή τους, ε, να βελτιώσουμε τους βοσκοτόπους, ε, να λάβουμε έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση, να, να επιδοτήσουμε τους γεωργού που οικειοθελώς μειώνουν την παραγωγή τους, ε, Επίσης να εφαρμόσουμε αποσύρσεις, ε, να αυξήσουμε την ιδιωτική αποθεματοποίηση, οποιαδήποτε μορφή στρατηγικής στήριξης της παραγωγής. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα άρσης παροσορινά τουλάχιστον των ε, δασμών, ιδιαίτερα από συγκεκριμένες προελεύσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποια κάποια καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ε, είναι 30% οι παράγοντε παραγωγή ε, για το κόστο μια εκμετάλλευση. Μόνο έτσι θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το γαλακτοκομικό τομέα ε, την Κροατία. Τον περασμένο χρόνο 2.000 γαλακτοπαραγωγοί σταμάτησαν ε, τη δραστηριότητά τους εξαιτία έλλειψης ε, πρόσβασης σε ε, πιστώσεις. Επίσης έχει μειωθεί κατά, κατά 3 λεπτά του ευρώ η τιμή του γάλακτος. Η μέση τιμή είναι περίπου 20 λεπτά του ευρώ το λίτρο το γάλα. Ε, στην Κροατία. Η είσοδος Κροατίας ε, στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών και μάλιστα από μεγάλες αλήθειες παραγωγής σε τιμές dumping. επιπλέον είχαμε το ρωσικό εμπάρκο και την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Στην Ευρώπη αυξήθηκε η γαλακτοπαραγωγή, ενώ στην Κροατία η παραγωγή γάλακτος μειώθηκε κατά 5% πέρυσι. Και επιπλέον οι γαλακτοπαραγωγοί στην Κροατία δεν έχουν που να διαθέσουν το γάλα, το γάλα τους εξαιτία του αθέμητου ανταγωνισμού. Τελικά καταλήγει στην λιγότερο προστατευμένη αγορά το γάλα τους, δηλαδή στην κροατική αγορά στην εγχώρια αγορά. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτησή μου. Τι εθνικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η Κροατία για να προστατεύσει τους γεωργούς της, τους κτηνοτρόφους της και επίσης ε, πιστεύετε θα πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα των αθέμετων εμπορικών πρακτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Αναμφίβολα θα πρέπει να λάβουμε μέτρα στην Ευρώπη. Διαφορετικά οι διακοιμάνσει αυτές των τιμών θα καταστρέψουν τελικά τους ίδιου του γεωργού και τους ίδιου τους κοινοτρόφου. Η κατάσταση λοιπόν όπως βλέπετε κύριε Επίτροπε είναι πάρα πολύ δυσχερής. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε τι το δυνατό για να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις. Το εμπάρκο της Ρωσίας όπως ξέρετε επηρέασε πάρα πολύ του Ευρωπαίου γεωργού και γνωρίζουμε επίση ότι Ακόμα και όταν ε, μειώνονται λίγο οι τιμές, ε, η επίπτωση είναι δεκαπλάσια για τους γεωργούς. Κύριε Πίτροπε, λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να δούμε τι είδου ενίσχυση μπορούμε να δώσουμε για του γεωργού εκείνου οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δεινή οικονομική κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να έχουμε νέε επενδύσει στο γεωργικό τομέα διότι γνωρίζετε κύριε Πίτρο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γεωργοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση απόγνωσης. Αυτούς ακριβώς τους γεωργούς πρέπει κατά προτεραιότητα να προστατεύσουμε και πρέπει παράλληλα να δούμε πώς θα καταφέρουμε να λάβουμε μέτρα πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με αυτή την ανάλυση κινδύνου που κάναμε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις κύριε Πίτροπε, κύριο ο Καταρχήν, για την κατάσταση στις αγορές ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιέρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο στη στήριξη αυτών των αγορών. Αλλά ακούσαμε και από εσά ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δραματική στην κατάσταση στι αγορέ γάλακτο σε όλα τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά την αγορά κρέατο. Ε, διαρωτώ με αν τα μέσα που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτελεσματικά. Γιατί πολλά χρήματα αφιερώθηκαν, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για την ολοκλήρωση ε, των ε, διαπραγματεύσεων των συνομιλιών με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε κύριε Επίτροπε ότι το θέμα των γεωργικών ενδείξεων ε, των εισαγόμενων προϊόντων από τις Ηνωμένε Πολιτείε ή η σήμανση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε προϊόντα των ΗΠΑ θα είναι ζητήματα που θα αποτελέσουν κόκκινες γραμμές και που δεν θα ενδώσει στις διαπραγματεύσεις τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα κάνει καμία απολύτως υποχώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε αριθμητικά στοιχεία ε, για τις ζημίες που έχουμε υποστεί από το εμπάργκο της Ρωσίας. Οι Γεωργοί πιστεύω ότι είναι τα πρώτα θύματα αυτού του εμπάργκου και πρέπει ε, να λάβετε περισσότερα μέτρα ε, από ό,τι αυτά τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική. Χαίρομαι που επιτέλους αναγνωρίζετε ότι είναι δραματική η κατάσταση διότι έχετε χάσει πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σα το έχουμε επισημάνει πολλέ φορέ, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατόν. Δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο στον προβληματισμό. Πρέπει να περάσουμε στη δράση. Ε, υπενθυμίζω ότι οι τιμές παρέμβασης καθορίστηκαν το 2008 και έκτοτε αυξήθηκαν κάποια έξοδα, κάποιες δαπάνες των αγροτών και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αγοραστική δύναμη σε πολλά κράτη-μέλη. Ακόμη, ε, το θέμα της επισήμανσης ε, των, του συστατικών κρέατος σε κάποια έτοιμα φαγητά σε κάποιες χώρες πρέπει να μας απασχολήσει και ε, το θέμα των αθέμητων πρακτικών όπως ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι. Ετοιμάζω μάλιστα και μια έκθεση για την αστάθεια των τιμών και θα με υποστηρίξουν και άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Κύριε Ράνς Καρσία. Κύριε Επίτροπε, είναι ελάχιστα πενιχρά τα αποτελέσματα του γαλακτοκομικού πακέτου. Είπατε να το διαβρύνετε, ε, να διαβρύνετε συμβατικές σχέσεις και σε άλλους κρίκους αλυσίτους, όχι μόνο στην πρώτη. Ε, προσωρινά να αυξήσετε τις τιμές παρέμβασης, έστω και προσωρινά. Επίσης, γιατί δεν χρησιμοποιείτε το άρθρο 222 της κοινή οργάνωσης αγορών, μετά την τελευταία μεταρρυθμίση που επιτρέπει στους ε, ε, συνεταιρισμού στο γεωργό στις οργανώσεις, στι δοκλαδικές οργανώσει, για έξι μήνε να αναλάβουν δράσει σε ό,τι αφορά την απόδοση των τιμών. Έτσι τουλάχιστον εξασφαλίστε μια αυτονομία τη διαχείριση για να βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεση τη νέα διατάξει, νέου μηχανισμού στην κοινή οργάνωση αγορά. Γιατί δεν του χρησιμοποιεί. Επιτέλου, χρησιμοποιήστε αυτού του μηχανισμού. Η κυρία Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πιο εντυπωσιακή δήλωση που έγινε σήμερα ήταν αυτή η τήρηση ενός λεπτού σιγής από τον κύριο Μποβέ. Γιατί πραγματικά κάτι πάρα πολύ σάπιο αυτή τη στιγμή βλέπω στη δική μας την κοινωνία, αν αυτοί οι οποίοι παράγουν τρόφιμα είναι τόσο τελικά απεγνωσμένοι που καταλήγουν τελικά στην αυτοκτονία. Και δεν είναι γαλλικό μόνο το φαινόμενο αυτό, σας διαβεβαιώ. Πρέπει λοιπόν να ρωτηθούμε πραγματικά πού ζούμε και τι κάνουμε όταν καταναλώνουμε εμεί τρόφιμα τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα από ανθρώπους που τα παράγουν και οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Βραχυπρόθεσμα, αυτό είπατε. Καλά κατάλαβα. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε πότε επιτέλου θα αναλευθεί δράση η οποία θα έχει πραγματικέ αποτελεσματικέ επιπτώσει. Γιατί ξέρετε ότι και ο σκληρό σύτο και τα προκυπευτικά είναι προϊόντα τα οποία έχουν πληγεί πέρα από τον τομέα του χείριου κρέατο ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και δεν μου έκανε καθόλου θετική εντύπωση η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί τι πίεση ασκείται αυτή τη στιγμή εσεί προκειμένου να γίνουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη διατροφική αλυσίδα. Κύριε αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε τον Επίτροπο ε, και ο όρος Επίτροπος είχε χρησιμοποιηθεί και στο ανώτατο Σοβιέτ. Κύριε Επίτροπε, δεν με πείσατε. Νομίζω ότι δεν απαντήσατε σε αυτά τα οποία περιμένουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Ε, είστε ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων στον αγροτροφημικό τομέα. Εμένα με ενδιαφέρει το θέμα του ανατάτου επίπεδου εγγύσεων που μπορούν οι κυβερνήσεις να δίνουν στους αγρότες. Δεύτερον, με ενδιαφέρει η εσωτερική κατανάλωση και η υποχρεωτική σήμανση την οποία αναμένουμε. Και επίσης η αύξηση των τιμών αναφοράς για το γάλα και για το χείριο κρέα γιατί είναι πολύ χαμηλή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι σαφές ότι χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, χωρίς επιπλέον ενισχύσεις, δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ή λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κονδύλια στο κοινοτικό προπολογισμό ή να ρυθμίσουμε τις τιμές. Αλλιώ η κατάσταση θα μείνει αμετάβλητη. Ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα. Ή τουλάχιστον να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τους γεωργούς να τους επιδοτήσουν. Η κατάσταση σε πολλά κράτη είναι κρίσιμη, στις βαλτικέ χώρε συγκεκριμένα, στη Λιθουανία. Εισάγουμε γαλακτοκομικά, κυρίως γάλα, από άλλε χώρες και οι τιμέ γάλακτο έχουν καταβαραθρωθεί. Οι κτηνοτρόφοι δεν θέλουν πια να παράγουν γάλα και σκέφτονται να αφήσουν τις αγελάδες τους μπροστά στη Λιθουανική Βουλή ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Έχουν ε, ήδη οργανώσει τέτοιες διαδηλώσεις ε, και θα πρέπει κάτι να κάνουμε και να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ο κύριος Τάκολα, Τάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Θα είμαι λακωνικότατος γιατί γνωρίζω ότι ξέρετε και εσείς ότι η κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα στη Φιλανδία είναι πολύ κρίσιμη και επιδεινώθηκε και με το ρωσικό εμπάργο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει και μάλιστα να βαθμίσει τη στήριξή της προς το γαλακτοκομικό τομέα. Θα πρέπει να προτείνετε μάλιστα και μέτρα να ε, περιορίσετε την παραγωγή γάλακτος στην ενιαία αγορά τώρα. Γιατί ένα από τα προβλήματα, τα προβλήματα της κατάργησης των γαλακτοκομικών προσωστώσεων είναι πια ορατά. Ερωτώ λοιπόν, Πρόκειται να προτείνετε μείωση της παραγωγής του γάλακτος στην ενιαία αγορά και να αυξήσετε το επίπεδο στήριξης στον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα. Ευχαριστώ κύριε Χόιμπους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι για δύο χρόνια θα διαθέσετε 900 εκατομμύρια. Στη Γερμανία και μόνος το γαλακτοκομικό τομέα και μόνο το 2015 είχαμε 3,2 δισεκατομμύρια ε, λιγότερα από τα απαιτούμενα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των αγροτών. Αυτό ίσως οφείλεται στις ε, εξαγωγές, αλλά οι εξαγωγές ε, των γαλακτοκομείων μπορούμε να πούμε ότι αυξήθηκαν το 2015. Οι τιμές εκτός από μόνο στο γάλα έμειναν σταθερές τα γαλακτοκομεία δείχνουν να έχουν έσοδα, να έχουν βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία, αλλά όχι ε, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Φαίνεται ότι ε, τα έσοδα τους μειώνονται. Φαίνεται ότι εξυπηρετούνται κάποια οικονομικά συμφέροντα, αλλά όχι τα συμφέροντα των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Ευχαριστώ. Πόσο Τζουφίλα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζουφίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Σας ευχαριστώ επίσης για, τα, για όσα μας είπατε. Πέρα από τις δηλώσεις που ακούσαμε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει πλέον ότι η κρίση αυτή είναι πάρα πολύ βαθιά και ιδιαίτερα ευρεία, διάχυτη θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε. Αναφερθήκαμε στην κρίση του γάλακτος, αλλά όχι στην κρίση της ντομάτας, ιδίως στις νότιες χώρες της Ευρώπης. Ιδίως σε κάποιες περιοχές της νότιας λοιπόν Ευρώπης. Ξέρετε ότι οι οργανώσεις παραγωγές μας έχουν πει ότι στις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου οι εξαγωγές από το Μαρόκο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν πάνω από 65%. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε σε πάρα πολύ σημαντική μείωση των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω στι νότιε αγορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τα δεδομένα αυτά και θα ήταν σε θέση να μα δώσει συγκεκριμένα τελειωνιακά δεδομένα όσον αφορά τι εξαγωγέ από το Μαρόκο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση, εσεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακολουθείτε πραγματικά τι ε, ποσότητε που μα έρχονται από τρίτε χώρε γιατί πάντα αναφερόμαστε σε εκτιμήσεις οι οποίες είναι ανεπίσημες, σε στοιχεία τα οποία είναι ανεπίσημα. Και θα μπορούσατε εσείς μονομερός να αναλάβετε κάποια μέτρα διάσωσης ε, των προϊόντων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ δινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιες αγορές. Μήπως θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε κάποιους τελωνιακούς δασμούς. Ευχαριστώ κύριο Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να σας συγχαρώ γιατί γίνεστε όλο και πιο θαραλέος και επιτέλους αναγνωρίζετε πράγματα που ε, εδώ και χρόνια επισημαίνουμε, εδώ και χρόνια σας κρούμε τον κόδωνα το κίνδυνο για την κρίση. Επιτέλους ξυπνήσατε. Καλά ξυπνητούρια. Επίσης είπατε ότι οι κτηνοτρόφοι στη Ρουμανία έχουν λάβει χρήματα για να περιορίσουν τις δημίες τους. Όντως ε, τα έχουν λάβει, αλλά για μη μεταποιημένα προϊόντα στη Ρουμανία. Οπότε δεν ε, έχετε κάνει σωστά τα καθήκοντά σας, ε, κύριε Επίτροπε, γιατί φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε καν τα στοιχεία. Επίσης, αν αρθεί το ρωσικό εμπάργκο στο μέλλον, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει σχέδια ήταν τεράστιε οι ζημίε εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Έχουν γίνει κάποιε μελέτε ε, τη αγορά. για να αποτιμήσουμε αυτές τις ζημίες και να εφαρμόσουμε μία στρατηγική βιώσιμη σε περίπτωση που αρθεί το ρωσικό εμπάργο. Αν υπάρχει αυτή η στρατηγική, θα θέλω να μας την παρουσιάσετε για να μην έχουμε τις άρεστε εκπλήξεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είναι σημαντική για μας η παρουσία σας εδώ και η ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιούμε. Ε, φαίνεται ότι ακούσατε τι προβλήματα έχουμε στη Ρουμανία με τις κρατικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις και τι δύσκολη και κρίσιμη περίοδο διανύουν οι αγορές μας και είχαμε και επιδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Ε, δεν ξέρω αν ε, γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια σωστή μηχανοργάνωση ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κεντρικό σύστημα πληρωμών και επιδοτήσεων για να μην έχουμε διαφορές στις πληρωμές των επιχορηγήσεων και των ενισχύσεων προς τους γεωργούς. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα με τα αγροτεμάχια. Υπάρχει ένα κοινή γεδαφών και γεών γεωργικών στην Ρουμανία. 40% των γεών έχουν περάσει σε χέρια λαδαπών επενδυτών. Αυτό που μόνο δεν είναι πρόβλημα, αλλά μακάρι να χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς ε, αυτά τα εδάφη, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Ο κύριος Νούνο Μέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Δεν είστε τόσο πολλά χρόνια ε, επίτροπος για να είστε εσείς ε, ο έρον όλα τη αμαρτίε του κόσμου και ο υπεύθυνο όλων των κακών τη κοινή γεωργική πολιτική. Απλώ προσπαθούμε να βρούμε από κοινού λύσει. Και το θέμα δεν είναι ε, να πληρώνουμε κάποιον για να δουλέψει, αλλά να αποδίδει η γεωργική δραστηριότητα. Και καμία οικονομική δραστηριότητα δεν είναι δυνατή χωρί κέρδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαιτούμε από τους γεωργούς να έχουν γεωργική δραστηριότητα χωρίς κέρδος και να δουλεύουν ε, για την ψυχή τους. Γιατί ε, φαίνεται ότι με όλα τα μέτρα που προτείνουμε δεν έχουμε καμία πρόοδο και καμία αλλαγή. Και μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γιατί η Γεωργία εξασφαλίζει την επιστημιστική αυτάρκεια της Ευρώπης, εξασφαλίζει θέσεις απασχόλησης, η Γεωργία εξασφαλίζει μια σωστή χωροταξία αλλά δυστυχώ δεν εξασφαλίζει γεωργικό εισόδημα για όλου του γεωργού. Είχαμε γαλακτοκομικέ ποσοστώσει, καταργήθηκαν. Έπρεπε να βρούμε μια λύση. Η λύση ήταν ναι, η ποσοστό για ένα διάστημα, αλλά οι ποσοστώσει καταργήθηκαν. Επίση έγινε άνοιγμα των αγορών ε, προ άλλε αγορέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που μα κατακλείζουν με προϊόντα σε τιμέ dumping. Με αποτέλεσμα να καταβαραθρώνονται, να καταραίουν οι τιμέ στην Ευρώπη. Δύο ερωτήσει. Για το ρωσικό εμπάργο. Πρόκειται επιτέλου να αρθεί. Δεύτερον, τι γίνεται με το TTIP και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είμαι κατά του TTIP, αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε κάποιε ασφαλιστικές δικλείδες για τους γεωργού μα παρακαλώ, στο TTIP. Ο κύριος Νταντά. Κύριε Πίτροπε, Καταρχά σα ζητώ συγγνώμη Συγγνώμη γιατί τη η πτήση μου και δεν μπόρεσα να ακούσω την αρχή σας παρέμβαση. Μου είπανε πάντως πολύ πιστά τι είπατε. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, για πολλές μέρες είχα πάει στην έκθεση αγροτικών προϊόντων που γίνεται στο Παρίσι και αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά εντύπωση ήταν η εγανάκτηση και η οργή των ε, γεωργών. Ακόμα και αυτοί που θεωρούν ότι είναι η καλύτερη παραγωγή γάλακτος, ε, κρέατος κτλ. Ακόμα και οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δινή θέση. Σε μια προηγούμενη συνεδρίαση μας είχατε πει ότι οι δείκτες αυτή τη στιγμή δεν αποδεικνύουν ακόμα το φαινόμενο αυτό. Να σας πω όμως εγώ, να σα δώσω εγώ κάποιου δείκτες κύριε Επίτροπε, γιατί μπόρεσα να ακούσω τους ε, γεωργού. Ένα 15% των γεωργικών των σε ορισμένες περιοχές δεν αποδίδουν πλέον χρήματα. Επίσης, η κατά 40% έχουν αυξηθεί τα τέλη τα οποία βαρύνουν τους γεωργούς σε σχέση με την περίοδο την ίδια πέρυσι. Όταν συζητούμε με τους βιομήχανους μας λένε ότι έχουν χάσει 14% στην τιμή του γάλακτος, 30% από το περιθώριό τους και στην εβδομάδα μετά το τέλος διαπραγματεύσεων, ορισμένοι είδανε ότι χάσανε περίπου 30 προϊόντα. Αυτά στις διαπραγματεύσεις που έχουν αυτοί οι βιομήχανοι οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού κλάδου με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο βλέπετε ότι δεν καταφέρουν να πληρωθούν και οι ίδιοι γεωργοί. Στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προβάλει πολύ περισσότερε και πιο μεγαλεπίβολε προσδοκίε. Είχαμε πει τότε ότι σε περίοδο κρίση θα πρέπει οι οργανώσει των παραγωγών, καθώ επίση και σχετικοί του σύλλογοι, να μπορούν να παρεκκλίνουν από το 201 παράγραφος 1 της συνθήκης, δηλαδή το άρθρο εκείνο το οποίο ρυθμίζει το δίκαιο του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση στις υφιστάμενες διαπραγματεύσεις να ευνοήσουμε και να ενισχύσουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέση των γεωργών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο ελπιδοφόρη η κατάσταση. Και αν δεν κάνω λάθος κύριε Πρόεδρο, όσον αφορά δύο στις εξαγωγές, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα πόλεμο τιμών, όπως είπε ο κύριος Ταραμπέλα πριν από λίγο. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά προϊόντα να συνοδεύονται από καλύτερα συστήματα προώθησης, προκειμένου να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Αν δεν καταφέρουμε γρήγορα να κάμψουμε, η απόγνωση είναι τέτοια αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο, που νομίζω πραγματικά θα καταφέρουμε ποτέ να ανακάμψουμε από την κρίση αυτή. διπλα, σας άφησα διπλάσιο χρόνο ε, γιατί εσείς ε, ήσταν ο εμπνευστής ε, αυτής της συνάντησης, της έκτακτης συνεδρίασης και νομίζω ότι η δυναμική των λαγών είναι έκτακτη αυτή τη στιγμή. Είναι εξαιρετικού χαρακτήρα και η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν πήγε προς την επιθυμητή κατεύθυνση αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό και είναι έκτακτη αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε κάποιες δράσεις για να διορθώσουμε τη ερώτα μας και μετά να δούμε και ποιες είναι οι συστημικές αλλαγές που χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για να δούμε τι γίνεται και σήμερα αλλά και τι θα γίνει μετά το 2020 έχουμε το εδώ και τώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές ανάγκες και αργότερα να δούμε ποιες συστημικές αλλαγές θα χρειαστούν. Πάντως οι τιμές των, των γεωργικών προϊόντων παγκοσμίω ε, μειώνονται, μειώθηκαν τον περασμένο χρόνο ε, και λόγω της ε, αύξησης της ζήτησης, αλλά και η αύξηση της παραγωγής, της κατανάλωσης ε, ή μάλλον τις μείωσης συγγνώμη της κατανάλωσης, γιατί λένε ότι η λακτόζη τη μία το κατανάλωση, επίσης ε, είναι βλαβερό, μειώνεται η κατανάλωση. κρεα επίση ειναι βλαβερο μειωνεται επηρεάζει οι αλλαγέ στην ε, ε, ζήτηση, επηρεάζει και την κατάσταση των γεωργών και την προσφορά. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, το ποσοστό γενικώ, αλλά ε, πολλοί μιλούν για τις συμβάσεις. Ε, οι συμβάσεις δεν είναι μια σύγχρονη μορφή ποσοστώσεων σε τελική ανάλυση. Επίσης, τι γίνεται με το εμπάργο. Θα αλλάξει η κατάσταση. Ε, τι γίνεται η κατάσταση της ρωσικής γεωργίας που γίνεται όλο και πιο αυτάρκης, οπότε δεν θα χρειάζεται τόσες πολλές εισαγωγές προϊόντων. Κύριε Επίτροπε, έχετε 15 λεπτά και ευχαριστώ και τον περαιτέρω τους διερμηνείς για την παράδοση του ωραρίου. Ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις έκανα μια-δυο προτάσεις, αλλά βέβαια αυτά που είπα στην αρχή δεν είναι όλα τα μέτρα τα οποία προτείνεται να παρουσιάσει η Επιτροπή. Είναι περιορισμένοι η πόροι μας, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μέσα σε περιορισμένους πόρους δουλεύουμε και περιοριζόμαστε και από την νομοθεσία. Με τα εργαλεία που έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και προσπαθώ να έχω και υποστήριξη από τους άλλους επιτρόπους. Και βεβαίως ε, και ο ανταγωνισμό παίζει ρόλο. Έχει δίκιο και ο κύριος ε, Νταντάν και οι άλλοι συνάδελφοι. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού βλέπει διαφορετικά τα πράγματα από ότι πολλοί από εμά ε, στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και μπορείτε να αναμένετε ισχυρέ αντιστάσεις από άλλες γενικέ διευθύνσει όπω του ανταγωνισμού. Συνοψίζοντα όμω τα βασικά θέματα γιατί ε, μόνο τα βασικά θέματα μπορούμε να συνοψίσουμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Η ρύθμιση ε, της ε, παραγωγής και το άρθρο 222 αναφέρθηκε από πολλούς και είμαι πρόθυμος να το εξετάσω αυτό το θέμα. Το άρθρο 222 το έχουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού επ' αυτού. Εάν οι ενώσει παραγωγών και οι συνεταιρισμοί θέλουν ε, να λάβουν δράση για να προσπαθήσουν να ρυθμίσουν την παραγωγή, θα μπορούσαν να καλύψουν το 15% της παραγωγής γάλακτος και όχι το σύνολο της παραγωγής. Είναι μια εθελοντική ε, ρύθμιση και θα πρέπει να καλύψει αυτούς οι οποίοι το επιθυμούν σε κάποια κράτη-μέλη και μπορεί να μην έχει καμία επίπτωση σε άλλες χώρες όπου θα θέλουν να συνεχίσουν την παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 παρήγαγε 2,5% περισσότερο γάλα και οι τιμές ε, ήταν ε, σε κακή κατάσταση και ε, έβαιναν μειούμενες. Υπάρχει λοιπόν μείωση της τιμής και παράλληλα αύξηση της παραγωγής. Η τάση των τιμών δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στην παραγωγή. Πάντως εξετάζουμε τις δυνατότητες θελούσιας ρύθμισης της παραγωγής και με βάση το άρθρο 222 και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούν να εγκριθούν κάποια μέτρα σε αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε επίσης η παρέμβαση. Ε, και ο λόγο για τον οποίο έχω αντίρρηση είναι ότι αυτό δίνει άλλη μία διέξοδο για αυτού που θέλουν να παράγουν περισσότερο. Δεν περιορίζει λοιπόν την παραγωγή, πάει ακριβώς αντίθετα από αυτό το οποίο λέτε εσείς ε, για τη μείωση της παραγωγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα αν ε, το κάνουμε ελκυστικό και τους δίνουμε άλλη μια διέξοδο εκτός από τις χώρες ε, ε, του τρίτου κόσμου, αλλά, των τρίτων χωρών, συγγνώμη, αλλά τους δίνουμε και, την, και αυτό το μέτρο, θα, παράγουν περισσότερο. Αυτή είναι η, η πραγματικότητα. Θα μας κοστίσει και χρήματα παράλληλα, αλλά θα έχει και αρνητική επίπτωση στην πολιτική που να επιτύχουμε, του να περιορίσουμε την παραγωγή αν Αναφέρθηκαν οι 190.000 ε, ε, τόνοι όσον αφορά την παρέμβαση. Δεν νομίζω ότι ε, καλύπτεται το κενό. Θα πρέπει να βάλουμε ένα δίκτυο ασφαλείας σε ελκυστικές σημαίες και προσπαθούμε να έχουμε τα μέτρα τα οποία δεν θα αφήσουν τις τιμές να, να μειωθούν. Εξετάζουμε λοιπόν ε, στις υπηρεσίες της Επιτροπής τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε τα ανώτατα όρια και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση σε σχέση με το δίκτυο ασφαλείας για την παρέμβαση. Είμαι λοιπόν θετικά διατεθειμένος να το εξετάσουμε. Αναφέρθηκαν και τα οικονομικά στοιχεία και ο κύριος Ντές και άλλοι ανέφεραν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, ή ε, και άλλων ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναφέρθηκε και ε, το σχέδιο Juncker παράλληλα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να εξετάσει το θέμα βλέποντας και ε, τους κινδύνους που υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για αναδιάθρωση του χρέου των αγροτών για να μπορέσουν να, να ε, χρειάζονται ειδικά μέτρα που διανύουμε ειδικέ περιόδους ε, κρίσης. Θα δούμε μήπως μπορούν να διαμορφωθούν νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Το κόστος εισρώων τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και η αγορά λιπασμάτων ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Είναι δύσκολο ε, να ανταγωνιστούν λοιπάσματα άλλων χωρών, τα ευρωπαϊκά λοιπάσματα, με το τωρινό δασμολογικό καθεστώς. Και με τον Επίτροπο Μοσκοβισή έχουμε συζητήσει το τι μπορεί να γίνει για μια προσωρινή αναστολή των δασμών ε, για τις τιμές των λοιπασμάτων. Αυτό θα είχε άμεση επίπτωση στο κόστος εισρώων ε, για τους γεωργούς. Ε, αν μπορούσαμε να επιτύχουμε μια μείωση 14 ευρώ ανά θα ήταν τεράστια η επίπτωση. Γιατί αυτή τη στιγμή το κόστος εισρώων δεν έχει μειωθεί όσο έχει μειωθεί αναλογικά η τιμή της ενέργειας. Θα εξετάσουμε λοιπόν και αυτό το κομμάτι της εξίσωσης για να μπορέσουν να έχουν καλύτερο περιθώριο κέρδους και κερδοφορίας οι αγρότες. Ενίσχυση ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χείριο κρέα είναι το άλλο θέμα. Πέρυσι είχαμε δύο τέτοια καθεστώτα με κόστος 44 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά κάποια κράτη-μέλη δεν συμμετέσχουν η Γαλλία συγκεκριμένα, όπου 2,5 εκατομμύρια τόνοι από τα 19 εκατομμύρια τόνων συμμετέσχουν μόνο. Οι εμπορευόμενοι δεν συμμετέσχουν για λόγους χρηματορών. Εμείς όμως προσπαθήσαμε ε, να το κάνουμε ε, ε, προς χάρη των παραγωγών. Η Γερμανία και η Ισπανία συμμετέσχουν με 25 εκατομμύρια τόνους σε κάθε χώρα. Λειτουργήσε σε κάποιες χώρες, λειτουργήσε στην Πολωνία, δεν λειτουργήσε στη Γαλλία, δεν λειτουργήσε στη Ρουμανία ήταν απογοητευτική η συμμετοχή σε αυτές τις χώρε. Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη αποδοχή του μέτρου. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τι θα είναι ελκυστικό στο μέλλον ως μέτρο. Βεβαίως όμως και είναι υπό εξέταση ο τομέας του χειρίου κρέατος. Δεν είχαμε την βελτίωση των τιμών που θα θέλαμε να δούμε ε, με, τον, ε, με την ποσότητα που βγήκε από την αγορά. Θα πρέπει να βρούμε τον προπολογισμό για να μπορέσουμε να έχουμε άλλο ένα καθεστώς ε, το, αντίστοιχο το 2016. Αν δεν αυξηθούν οι τιμές όπως ελπίζουμε, κάτι θα πρέπει να κάνουμε τους επόμενους μήνες. Και πάλι κάποιο ρόλο μπορούν να παίξουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι φορείς για την αναδιάθρωση του χρέους. Τώρα για τα διαθέσιμα μέσα. Είπε η κυρία Μαγκίνες ότι υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. και τα κράτη-μέλη μπορούν να μεταφέρουν χρήματα από ένα μέτρο ανάπτυξης της σε ένα άλλο μέτρο ανάπτυξης υπαίθρου μπορούσαμε να έχουμε τέτοια μετακίνηση από το ένα μέτρο στο άλλο μέσα σε έξι μήνες, τώρα μπορούμε να το έχουμε σε, μεγαλύτερο, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε αιτήματα των κρατών μελών, ε, ε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους δώσει ευελιξία για τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται υποπίεση σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αν διαβάσετε τον κατάλογο των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, υπάρχουν θέματα σταθεροποίησης του εισοδήματος, ασφάλειας. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία δεν χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Κατά μέσο όρο, η χρήση των εργαλείων που είναι διαθέσιμα, εργαλεία τα οποία εσείς έχετε δώσει, μέσω της νομοθεσίας που ψηφίσατε, θα δείτε ότι 7 από τα 19 μέτρα έχουν χρησιμοποιηθεί. Άρα θα μπορούσε η Επιτροπή σας να εξετάσει πώς μπορούν αυτά τα μέτρα να γίνουν πιο ελκυστικά για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες που τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά τη στοχευμένη ενίσχυση, 10 από τα 28 κράτη-μέλη μόνο ζήτησαν αυτά τα μέτρα τα οποία ψηφίσαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Όταν τα χρήματα τα οποία δώσαμε δεν δαπανώνται από τα κράτη-μέλη, είναι δύσκολο να επανέλθω εγώ με νέε προτάσει προ αυτήν την κατεύθυνση, που βλέπω ότι δεν απορροφώνται αυτά τα κονδύλια. Φαίνεται ότι η απορρόφηση είναι πολύ μικρή. Υπήρχαν πολλά χρήματα, τα 420 εκατομμύρια ήταν μεγάλο ε, κονδύλι, αλλά τα κράτη-μέλη δεν επωφελήθηκαν, επομένω δεν επωφελήθηκαν αντίστοιχα και οι, αγρότες, και οι αγρότες. Όλα αυτά λοιπόν ε, είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν με τα κράτη-μέλη. Τώρα η κατάσταση με τη Ρωσία. Κανεί από εμά στην αίθουσα αυτή δεν δημιουργήσαμε την κατάσταση, αλλά εμεί πρέπει να υποστούμε τι ε, ατυχεί συνέπειε είναι αποφάσεις ε, πολιτικές, αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και θα θέλαμε να εξομαλυνθούν οι εμπορικές σχέσεις, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Εγώ οφείλω να συνεχίσω να δίνω χρήματα στα κράτη-μέλη, να υποστηρίζω ε, τους τομείς που επλήγησαν από το εμπάρκο της Ρωσίας. Και αναφέρθηκαν σημαντικά ε, σχόλια ότι όταν ο Υπουργό Γεωργία τη Ρωσία είναι σε ένα κατάλογο ανεπιθύμητων προσώπων και δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να κάνουμε διαπραγματεύσει μαζί του. Ελπίζω να μπορέσουν ε, κάποια μέτρα να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις και ε, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Εσείς θα μπορούσατε ίσως να μιλήσετε με ε, τους Υπουργούς Εξωτερικών για να μπορέσουν να εξομαλυνθούν και οι εμπορικές σχέσεις. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ σε κάθε ευκαιρία και τονίζω το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Για μας δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Αν με ρωτάτε πότε θα λήξει αυτή η κατάσταση, η απάντησή μου είναι δεν ξέρω. Γιατί οι ανώτεροι μου αποφασίζουν και ξέρω ότι ο πρόεδρο Γιούγκερ θα ήθελε να βοηθήσει και κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει, αλλά το ταγκό χρειάζεται δύο για να, το χορέψουν και δεν ξέρω αν υπάρχει προθυμία και από τι δύο Αναφέρθηκε και το θέμα του de minimis, το οποίο εξετάζουμε. Όταν ανέφερε εγώ τις εξαγωγικέ πιστώσει, εννοούσα την, δυνατότητα των κρατών μελών να εξάγουν προ τρίτε χώρες. Όχι ε, επί τη βάση των αποφάσεων του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι, γιατί ε, στις διαπραγματεύσεις εκείνες προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες και δεν υπαναχωρούμε ως προς αυτό, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για εξαγωγικές εγγύησεις που μπορούν να δοθούν για ευαίσθητες αγορές, ούτως ώστε οι εμπορευόμενοι να μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους και βεβαίως και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε dumping, αυτό δεν θα μας το επέτρεπαν οι κανονισμοί του ΠΟΕ και δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός εγγύησης των εξαγωγών που έχουν χρησιμοποιήσει η Γερμανία και 13 κράτη-μέλη και εξετάζουμε κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει περισσότερο ευχρηστός για να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν βεβαίως για την ε, εφοδιαστική αλυσίδα και το ανέφερε η κυρία Μαγκίνες αλλά και άλλοι βουλευτές είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η τιμή του γάλακτος στη Γαλλία μειώθηκε ένα λεπτό του ευρώ αναλύτρο τους τελευταίους μήνες κατά μέσο όρο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που φτάνει στους ε, αγρότες και ανέφερε τη Γαλλία ως παράδειγμα. Στις περισσότερες χώρες συμβαίνει αυτό, στα περισσότερα κράτη-μέλη αυτό το οποίο γίνεται στην ε, λυσίδα παραγωγής δεν έχει επιπτώσεις στον παραγωγό. Και θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω και με την κυρία Βιενκόφσκα θα το, το, συζητήσω το θέμα αυτό, το συζητώ συνεχώς και θα συνεχίσω να το συζητώ και μπορεί και εκείνη να έρθει στην Επιτροπή σας για να το συζητήσετε, διότι το περιθώριο κέρδους ε, των αγροτών δεν μπορεί να μειώνεται κάθε χρόνο. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Εγώ είμαι λοιπόν υπέρμαχος αυτών των προτάσεων και στην Task Force για την Γεωργία και την Αγορά εξετάζεται το θέμα αυτό για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν χρειάζεται, εγώ είμαι ανοιχτό και θα το προωθήσω. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αλλά ας δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό το οποίο και εμείς και άλλες γενικές διευθύνσεις θα αποφασίσουν ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συγκεκριμένα. Με συγκίνησε πολύ η παρέμβαση του κυρίου Μποβέ. Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος της αγροτιάς. Μην νομίζετε ότι δεν είμαι ευαίσθητος ε, στην ε, δυστυχία των ε, αγροτών. και χρήματα έχουν δοθεί και δισεκατομμύρια έχουν δοθεί για τους πρόσφυγες και είναι δύσκολο να βρούμε χρήματα και ως Επίτροπος δυσκολευόμαστε. Ως Επίτροποι δυσκολευόμαστε να βρούμε κονδύλια για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας αυτές τις δύσκολες εποχές γιατί δεν θέλουμε να πλήττονται οι αγρότες, δεν θέλουμε να φύγεται η υγεία τους δεν περιμέναμε ότι η κρίση θα διαρκέσει τόσο πολύ και θα είχε τόσο σημαντικέ επιπτώσεις. Θα υποβάλουμε λοιπόν προτάσει την επόμενη εβδομάδα. Θα σκεφτώ πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Δεν ήθελα σήμερα να υποβάλω προτάσει, κύριε Πρόεδρε. απλώ μου δόθηκε η ευκαιρία να σα μιλήσω για την νομοθετική διαδικασία. Θέλαμε να μιλήσουμε και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο και την αρμόδια Επιτροπή Γεωργία. Και την επόμενη εβδομάδα θα παλέψουμε για το πακέτο μέτρων τα οποία θα θέλαμε να είναι πακέτα χρήσιμα για τους αγρότες και με τα νομοθετικά εργαλεία που θα προτείνουμε την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να προτείνουμε πόρους που θα είναι χρήσιμοι για τους αγρότες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, συλλογικά θα λάβει την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε είναι σημαντικό να συνομιλήσουμε με όλους τους επιτρόπους και να δούμε και τις σχέσεις με τις ε, χώρες μέλη για να επηρεάσουμε και τη θέση στο Συμβούλιο, αλλά να έχουμε συζητήσει και με τις πολιτικές ομάδες. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μεταφέρουμε σε όλα τα κατάλληλα πολιτικά επίπεδα και να προσετεριστούμε και άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές, να πείσουμε και τους αρχηγούς των ομάδων να δημιουργήσουν ένα πρόσφορο κλίμα ώστε να γίνει δεκτή η πρόταση του Επιτρόπου Χόγκαν. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί μόνο με συνεργασία θα καταφέρουμε ένα αποτέλεσμα που είναι σημαντικό, αναγκαίο και επιθυμητό από όλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε στη συνεδρία, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για το επιπλέον τέταρτο που μας παραχώρησαν. Μπορέσαμε όμως έτσι να διεκπαιρεώσουμε το έργο, και να, το έργο μας, τη συνεδρίασή μας και να ακούσουμε μέχρι τέλους τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ και εσάβρεν τα σπουδαία.